Uh, next point. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues, next point. Uh, Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι ψηφοφορίε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη σε όλους που χρειάστηκε να περιμένετε 15 λεπτά. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά είχαμε μια πολύ ζωηρή συζήτηση ως συντονιστές με πολύ καλά αποτελέσματα. Όλα βαίνουν καλώς, καμία ένταση, όπως βλέπετε μετά από τη συνεδρίαση, αλλά χρειαστήκαμε περισσότερο χρόνο από τον αναμενόμενο. Γι' αυτό ακριβώς υπήρξε καθυστέρηση, γιατί έπρεπε να τελειώσουμε με όλες μας τις δραστηριότητες. Τώρα λοιπόν έχουμε τέσσερις ψηφοφορίες, τέσσερις εκθέσεις και θα χρειαστούμε μια μισή, μια μισή ώρα Μία. Περισσότερα από μία ώρα. Να είσαστε έτοιμοι ψυχολογικά. Πάμε λοιπόν στην ε, έκθεση για τις ευρωπαϊκές στατιστικές για, τον, ε, για την ηλεκτρική ενέργεια, τη μόνο αερίου ηλεκτρικής ενέργειας. Μπάρμπαρα Κάπελ. Και καταρχήν κάνουμε μία δοκιμή. Καταρχήν ερώτηση, έχετε θυμώσει μαζί μας, γιατί καθυστερήσαμε, άρχεται η ψηφοφορία. Δοκιμή, δοκιμαστική. Πέρας. Ένας από το ΕΛΚ, ένας υπεράριθμος. Βλέπετε, γι' αυτό χρειάζεται η δοκιμαστική ψήφος. Γι' αυτό χρειάζεται ο έλεγχος. Κατάλογος ψηφοφοριό. Τροπολογία 68 μέχρι 56 με 68. Είναι παρόμοιες. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτονται. 73 και 76 on block υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 78 υπέρ 75 με συγχωρείτε υπέρ Against. κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οκτώ υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 80, 80, πέρας. Από το ΕΛ και το ΑΛΤΕ έχουμε έναν υπεράριθμο. Από το ΕΛΚ ακόμα Πέρας. Ωραία. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85. Ελέγχουμε την 85. Πέρας. Απορρίπτεται. 87, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε επί τις 88. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Επί της 89. Πέρα της ψηφοφορίας. Δεκτή. 90 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 90. Ψηφίζουμε επί της 90 ηλεκτρονικός. Πέρα ψηφορίας. Δεκτή. 91 μέχρι 61 τροπολογίες είναι ένα μπλοκ ψηφίζονται ομού. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 10 82-83 ομού οι τρεις αυτές υπέρ κατά δεκτές 84 υπέρ συγγνώμη συγγνώμη περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 20 Περάσαμε λοιπόν στην τροπολογία 20. Ψήφι Κατά. Ας επαληθεύσουμε την 20. Πέρα ψηφορίες. Απορρίπτεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα από την 21 μέχρι την 32 ομού ψήφι περ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107 και 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 μέχρι και την 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ Ας επαλθέψουμε την 40 παρατηρεί ο πρόεδρος επαλήθευση επί τη 40. Πέρα εφορία. Απορρίφθηκε. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικός άρχιρη ψηφοφορία επί του συνόλου της έκθεσης. Πέρας ...39 ψήφι υπέρ, 6 κατά. Έγινε δεκτή. Τώρα ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία και εδώ ηλεκτρονικό θα γίνει λοιπόν η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Και τώρα στην διαθεσμικές διαπραγματεύσεις χρειαζόμαστε την πλειοψηφία των ε, μελών της Επιτροπής, ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν, για τις ε, δύο οργανικές ε, διαπραγματεύσεις, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Υπάρχει λοιπόν συντριπτική πλειοψηφία. Εντάξει, έγινε δεκτή η εντολή για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή και με την κυρία εισηγητή, συγγνώμη. Περνάμε τώρα στην ε, επόμενη έκθεση για την ενεργειακή απόδοση. συγγνώμη, για την ε, ανανεώσιμη πηγές ενέργειας, ε, συμβαστική τροπολογία 13, ψήφι υπέρ, 59 υπέρ, κατά. Να σε επαληθεύσουμε. 59. Πέντε ψηφορίες. rejected oral. Basilikas, you should go for the card. Yeah. Rejected. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 14. Συμβαστική 14. Τι συνέβη, πάρετε και ο Πρόεδρος. You closed the vote too early. Βιαστήκατε να κλείσετε την ψηφοφορία, Πρόεδρε. Okay. okay? Okay. Okay. Uh, Συμβαστική 14. Όχι, όχι. Όχι, Πρόεδρε, όχι. όχι. Για την 59, την 59 για αυτή μιλάμε, στην οποία βιαστήκατε να κλείσετε την ψηφοφορία. Κύριε Πρόεδρε, Θέλετε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Μα δεν ψηφίσαμε την 59, διότι δύο μηχανήματάκια εδώ δεν δουλέψανε. Επαναλάβατε λοιπόν την ψηφοφορία διότι δύο συνάδελφοι δεν ψήφισαν. Το μηχάνημά τους δεν λειτουργούσε. You can, check. You have not two votes uh, Συνάδελφοι, εντάξει, θα χρειαστούμε δύο ώρες ε, για την ψηφοφορία, δεν έχω αντίρρηση αλλά εν μέσω της διαδικασίας δεν μπορούμε να αλλάζουμε τους κανόνες τον ίδιο χρόνο για την ψηφοφορία είχαμε για κάθε τροπολογία από μια στιγμή στην άλλη δεν μπορώ να αλλάξω εντάξει θα περιμένω περισσότερο χρόνο θα περιμένω περισσότερο χρόνο όταν είναι ονομαστική ψηφοφορία θα χρειαστούμε ίσως δύο ώρες εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα διότι πρέπει να είστε πεπισμένοι για το αποτέλεσμα της ψηφορίας. Λυπούμε, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε ψηφοφορία που έχει διεξαχθεί. Δεν υπήρχε κανένας ειδικό λόγος. Εντάξει, θα περιμένω περισσότερο χρόνο. Λυπάμαι για αυτό που συνέβη, αλλά δεν μπορώ να επανέλθω. Συμβαστική τροπολογία 14, ψήφι υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Συμβαστική 14. Θα περιμένω λοιπόν περισσότερο. Υπάρχουν ε, υπεράριθμοι στο ΕΛΚ, πέρα τη Δεκτή. Εντροπολογία. Η ε, προσθήκη στην 14 υπέρ, κατά. Επαλήθευση την προσθήκη στη συμβαστική 14. Επαλήθευση. Ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτή. 15 ε, τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτή. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε. 72. Ε, Έλεγχος επί της 72. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 18. Ε, 80, συγγνώμη. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 84 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. Συμβαστική 18. Έληξε ψηφορία. Απορρίπτεται. 92. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. 85 υπέρ. Κατά. Για μια ακόμα φορά, για την 85. Προπολογία 85. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να επαληθεύσουμε. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτή. Περνάμε στην 90. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. 90. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για μια ακόμα φορά. 91. Πέρα ψηφορίας. Απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 101. Ψήφι υπέρ. Κατά. επαληθεύουμε. 101. I close the vote. Πέρασε. Εκατόν δέκα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ρέτζι 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 123 υπέρ. 131 συγγνώμη υπέρ κατά. Θα επαληθεύσουμε 131. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα ψηφορίας. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. εποχές επαλήθευση. 132 τριάντα δύο. Πέρα Απορρίπτεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 137 ψήφι υπέρ κατά ας απελθέψουμε 137 πέρας δεκτή 139 υπέρ κατά Θα επαληθεύσουμε. 139. Πέρα της ευφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 24 συμβαστική υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε Συμβαστική 24. πέρευση οφορίας Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σας. 146 υπέρ. Κατά. θα επαληθεύσουμε. 146. Έληξη ψηφοφορία. Δεκτή. 147 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. 147. Πέρας ψηφοφορίας.

πέρα της εφορίας. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Πέρα της εφορίας. Απορρίπτεται. 151 υπέρ. κατά εποχές δεκτή 152 υπέρ κατά επαλήθευση έληξη ψηφοφορία απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές δεκτή 154 υπέρ κατά. Ας επαληθεύσουμε. 154. Έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ένβη 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε ψηφοφορία. Δεκτή. 162 ως προστίκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προστίκη στη συμβαστική τροπολογία 25 υπέρ κατά επαλήθευση συμπλήρωμα στην βασική τροπολογία 25 έγινε δεκτή 164 υπέρ κατά 164. Έλεγχος. Πέρα εφορία. Δεκτή. 165. Περ, κατά, αποχές, δεκτή. 166 περ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 26 πέρ κατά, αποχές δεκτή. Προσθήκη στην ε, τροπολογία 26, ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 172, συγγνώμη παρατηρεί ο Πρόεδρος, ως προσθήκη στην προσθήκη στην τροπολογία 26. Τροπολογία 186 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. 186 ε, τροπολογία. Έλεξη ψηφοφορία. Δεκτή. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 174 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 188 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε καλού κακού 188 πέρας Δεκτή. 189 <clears throat> υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Προστίκη στο 29 υπέρ. Κατά αποχή. Αποχές. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. προσθήκη στην ε, τροπολογία 30 υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε προσθήκη στην συμβαστική τροπολογία 30 πέρα ψηφορίας απορρίπτεται τροπολογία 200 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε Προπολογία 200. Πέρα ψηφοφορία. ...201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. 201. Θέλετε να ελέγξουμε, εντάξει. Ελέγχουμε τη 201. Πέρας. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. 202 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 203 υπέρ κατά, ελέγχουμε. Δεν έλεγξα τις αποχές, εν πάση 203. Αποδεκτή. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 205 υπέρ. Κατά αποχές 205 ελέγχουμε πέρας αποδεκτή 206 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή 207 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή 208 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή συμβασμός 31 υπέρ κατά αποχές αποδεκτός υπέρ κατά αποχές αποδεκτή 218 συμβασμός 32 υπέρ κατά αποχές αποδεκτός 219. Προσθήκη στο συμφωνισμό 32 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 219 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται αυτή τη φορά. 224 υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε και πάλι. 224. Πέρας. Απορρίπτεται. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, αποδεκτή. 226 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 226 ελέγχουμε. 226 πέρας. Απορρίπτεται. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 228 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 228 ελέγχουμε. 228. Πέρας. Απορρίπτεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Μάλλον έγινε αποδεκτή. 229. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Αποδεκτή. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε θεωρώ. Δεν είναι απόλυτα σαφές. 230. Πέρας. Απορρίπτεται. 231 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβασμός 33 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτός. 33α υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτός. Ε, ε, προσθήκη στο 33α υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτός. 240 υπέρ. Κατά αποχές, ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε καλύτερα. 240 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 241 υπέρ. Κατά αποχές αποδεκτή 243 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 244 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 245 υπέρ κατά αποχές, ελέγχουμε, ελέγχουμε καλύτερα, 245 ελέγχουμε, 245 ελέγχουμε, πέρας, αποδεκτή, 246 υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε καλύτερα. 246 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 247 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 247. 247. Πέρας. Δεκτή. Συμβασμός 34. 34 υπέρ. Πρόεδρε. Θα ήταν σκοπό να βλέπουμε τα αποτελέσματα στην οθόνη, γιατί εσείς είπατε δεκτή ή απορρίπτεται, αλλά δεν είδαμε τους αριθμούς. Θέλουμε να έχουμε εικόνα. συμπιφασμός 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. Τροπολογία 255 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. 257 υπέρ. Κατά αποχές, ας ελέγξουμε καλύτερα. 257. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 35 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 35. Συμβαστική πρόταση 35. Έλεγχος. Πέρας. Αποδεκτός. Ε, συμβαστική πρόταση 36 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 36. Ελέγχουμε τη συμβαστική πρόταση 36. Πέρας. Απορρίπτεται αυτή τη φορά. 265 και 266 από κοινού υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε, παρακαλώ. Τις δύο τροπολογίες τις ελέγχουμε. 265-266. Πέρας. Απορρίπτονται. 267 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε καλύτερα δεν είναι σίγουρο 267 267 ελέγχουμε πέρας αποδεκτή 268 α πάμε στην επόμενη συνεπώς 268 268 υπέρ Κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 268. Ελέγχουμε. Πέρασε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι συμβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει όπως με την προηγούμενη. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόβλημα με τη, μηχανή, με το μηχάνημα. Γιατί εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να αλλάξω, ε, να ψηφίσω δηλαδή, ε, πριν κλείσει. Ναι, αυτό είναι πρόβλημα. Αργεί το μηχάνημα. Δεν έκλεισα την ψηφοφορία για την 268. 268, 268. Θα ήθελα όμως να αλλάξετε θέση. Να αλλάξετε θέση αν έχετε πρόβλημα. Πάρτε την κάρτα σας και πηγαίνετε κάπου αλλού. Και θα θέλαμε ή να μας βοηθήσει η τεχνική υπηρεσία με αυτό το θέμα. Καθίστε κάπου αλλού. Εντάξει, συνάδελφε Ταμπουράνο, ελέγξατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίζουμε επί της 268. Ελέγχουμε για τη 268 και ψηφίζουμε ξανά. Πέρας. Απορρίπτεται. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε. 269 ελέγχουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 270 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Δεν σαφές το αποτέλεσμα. Πέρασε. Αποδεκτή. Συμβαστική πρόταση 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτή. Τροπολογία 275. Υπέρ. Κατά. Αποχές ας ελέγξουμε. 275. Ελέγχουμε. 275. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 38 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Είναι πολύ σημαντικός ο έλεγχος. Συμβαστική πρόταση 38. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 276 και 277 από κοινού υπέρ. Κατά. Μάλλον απορρίπτονται, αλλά σε ελέγξουμε καλύτερα. Ελέγχουμε για τις δύο τροπολογίες 276-277. Πέρας. Αποδεκτές. 281 υπέρ. 281 υπέρ. Α, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 282 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 283 υπέρ κατά αποχές έμβη MV5 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή συμβαστική πρόταση 39 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή τροπολογία 289 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή 290 υπέρ κατά, ας ελέγξουμε καλύτερα, 290 ελέγχουμε, 290, πέρας. Αποδεκτή 291 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται 292 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεκτή. 293 υπέρ κατά αποδεκτή 2,94 υπέρ κατά τώρα πρέπει να ελέγξουμε 2,94 ελέγχουμε παρακαλώ πέρας απορρίπτεται συμβασμό 40 υπέρ κατά αποχές δεκτός προσθήκη στη συμβαστική πρόταση 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 302 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 302. 302. Πέρας. Απορρίπτεται. Πω πω, λέει ο πρόεδρος. 303 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. 303 έλεγχος. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική πρόταση 41 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 307 υπέρ κατά ας ελέγξουμε 307 έλεγχος 307 πέρας δεκτή 308 υπέρ κατά η ίδια πλειοψηφία δεκτή 309 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 310 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 310 έλεγχος. 310. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 42. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Έμβη 22. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 320. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 322 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα. 322. 322. Πέρας. Δεκτή. 323 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 324 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 326 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 327 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 328 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή 330 υπέρ 328 θέλετε να ελέγξουμε εντάξει ευχαριστώ ελέγχουμε την 328 επανερχόμαστε στην 328 ε, έλεγχος πέρας απορρίπτεται 330 υπέρ κατά αποχές ε, δεκτή 332 υπέρ κατά αποχές δεκτή 333 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε 333 ελέγχουμε παρακαλώ πέρας Απορρίπτεται 334 υπέρ. Συμβάσμα 43 υπέρ. Κατά αποχές δεκτός 342 ε, υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 343 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 344 υπέρ κατά αποχές δεκτή 345 υπέρ κατά αποχές δεκτή MV 24 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή άγκρι 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή άγκρι 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή άγκρι 15 Α, με συγχωρείτε, 5 λέει ο πρόεδρος, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, συμβαστική πρόταση 1, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, 4 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, συμβαστική πρόταση 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, συμβαστική πρόταση 3 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή, συμβασμός 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτός 12 υπέρ κατά Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. Τροπολογία 12. Έλεγχος. 12 ελέγχουμε. Πέρασε. Δεκτή. 14 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά αποχές δεκτός συμβασμός, ε, συμβασμός 6 υπέρ, κατά αποχές δεκτός συμβασμός 7 υπέρ, κατά αποχές δεκτός, συμβαστική πρόταση 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, συμβασμός 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτός, συμβασμός 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτός Συμβασμό 11 υπέρ κατά αποχές δεκτός τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβασμός 12 υπέρ κατά ας ελέγξουμε συμβαστική πρόταση 12 ελέγχουμε Συμβασμός 12, συμβαστική πρόταση 12 ελέγξαμε. Πέρας. Δεκτή η πρόταση. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε καλύτερα. Τροπολογία 48. Για να είμαστε απόλυτα σίγουροι. 48. Πέρας. Απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά. Ας ελέγξουμε καλύτερα 51, 51. Πέρας. Δεκτή. 58. Τροπολογία 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, να σκόντε τα χέρια παρακαλώ για να βλέπω. Ας ελέγξουμε. 58 και θα ήθελα να φαίνονται τα χέρια σας. Σωστή ανάταση. Πέρας. Δεκτή αυτή τη φορά. Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την έκθεση όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική, ηλεκτρονικά και ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε και είναι και ονομαστική ψηφοφορία παράλληλα. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται 34 υπέρ, 30 κατά, καμία αποχή. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Καθόλου εύκολη αυτή η ψηφοφορία, αυτή η έκθεση. From, from, from Λυπούμε, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα το έργο μας. Περνάμε στην έκθεση Μάρκους Πίπερ σχετικά με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Αγαπητοί φίλοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βλέπω ότι πολλοί από εσά έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται, άρα δεν ενδιαφέρονται πρωί 26 πέρα, Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Και παρακαλώ καθίστε. Ελέγχουμε τη 46. Πέρα της εφορίας. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Σαράντα ένα. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά Αποχέ. απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε 47 από τα πρώτα να παρακαλώ καλό θα ήταν να ψηφίζετε Γκέρετ, Λόπες κλπ αν δεν ψηφίζετε χάνω την επαφή με το κόμμα σας με την ομάδα σας πέρα ψηφορίες απορρίπτεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά αποχές αποχές. Συμβαστική μείον 3 υπερ Υπέρ. Δεκτή. NB2 υπέρ. Κατά αποχές. NB2 ε, ελέγχουμε Πέρα ψηφοφορία. Δεκτή. Συμβαστική τρία υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συνάδελφοι από το ΕΛΚ, παρακαλώ, καλό θέλετε να ψηφίζετε. Ζητώ συγγνώμη που σας κάνω την παρατήρηση, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. δεκτή. Ένβη 41. Συγγνώμη. Ένβη 41. Πέρα ψηφορίας. Δεκτή. Συμβαστική 3α υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη συμβαστική 3α. Πέρα ψηφορίας. Δεκτή. Ένβη 42 υπέρ. Κατά εποχές ας επαληθεύσουμε NV42 πέρα οφορία. δεκτή συμβαστική 16α ε, υπέρ κατά Αποχές επαλήθευση 16α. Πέρα ψηφορίας. Δεκτή. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. 65. Πέρα ψηφορίας. Δεκτή. 68 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση και εδώ 68 Πέραση της ψηφοφορίας συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4α υπέρ κατά αποχές συμβαστική τροπολογία 4α επαληθεύουμε δεν είναι εύκολο να μαντέψουμε ένας παραπάνω από τους σοσιαλιστές δημοκράτες πέρα της Δεκτή. NV43 υπέρ κατά αποχές δεκτή NV10 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση πέρα εφορίας δεκτή Συμβαστική 4β υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Συμβαστική 4β. Πέρα ψηφορίας Δεκτή. Προπολογία 2.34 υπέρ. 2.32 συγγνώμη. Υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. Συνάδελφοι, τροπολογία NV49 θα πρέπει να ψηφιστεί ως προστίκη Και 50 καταπίπτει τώρα. 49 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Υπέρ τη 49. Έληξη ψηφοφορία. Έγινε δεκτή. 77 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές θα επαληθεύσουμε. 82. Πέρας. Δεκτή. 83 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε. άρχιν ψηφοφορία, ψηφοφορία. Ένας πλεονάζει από τους S&D. Κλείνει ψηφοφορία, δεκτή. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές δεκτός. Συμβασμός 6 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτός. Τροπολογία 99 υπέρ κατά θα επαληθεύσουμε. Πέρα ψηφορίας Απορρίπτεται. Ένβη 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 102 υπέρ κατά αποχές δεκτή 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή 104 υπέρ κατά αποχές δεκτή 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή συνδεσμός 7 υπέρ ε, 105 θέλετε να ελέγξουμε θα ελέγξουμε 105 ελέγχουμε 105 ψηφίζουμε για την 105 ηλεκτρονικός ε, Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 118 έως 121. Τέσσερις τροπολογίες μαζί. Ψήφι υπέρ κατά επαλήθευση και για τα τις τέσσερις τροπολογίες. Πέρα ψηφορίας απορρίπτεται. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 124 Επαληθεύουμε την 124 πέρα της Απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση επί της 123 πέρα ψηφορίας απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 128 υπέρ κατά Ας επαληθεύσουμε. 128. Ψηφίζουμε. Έλλειψη ψηφορία. Δεκτή. Περνάμε στην 136. Όχι, συμβαστική 9. Συμβαστική 9. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 149 υπέρ κατά αποχές δεκτή 150 υπέρ κατά αποχές 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 159 υπέρ κατά Κατόν πέντε πέρα ψηφοφορίας έγινε δεκτή. 154 δεύτερο τμήμα ψηφιπέρ κατά Επαληθεύουμε. 154 δεύτερο τμήμα. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ένβη 39 υπέρ. Κατά. Αποχέσεις δεκτή. Ένβη 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 184 υπέρ κατά σε επαληθεύσουμε ε, επί της 184 πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται μου φαίνεται 185 υπέρ υπέρ κατά αποχές 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 189 υπέρ συγγνώμη 192 ψηφίζουμε υπέρ της ψηφορίας απορρίπτεται 189 και 191 190 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές δεκτές συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές δεκτό 200 υπέρ κατά θα σε το πολύ 200 πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται. 205 υπέρ κατά αποχές δεκτή 202 υπέρ κατά αποχές δεκτή 203 υπέρ κατά σε παληθεύσουμε 203 Έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 204 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. 204. Έληξη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 206 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 14 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή 217 υπέρ κατά αποχές δεκτή 218 υπέρ Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 226 υπέρ. Κατά. Ας επαληθεύσουμε. 226. Επαληθεύσουμε.

κατά αποχές συγκρίνεται 235 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε 235 επαλήθευση και πέρας απερίφθη 236 υπέρ κατά Αποχές απερίφθη. Εγκρίνεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 238-239 μαζί. Ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. 238-239 από κοινού. Πέρας. Απερίφθη. 241 υπέρ. Κατά. Για άλλη μια φορά επαληθεύουμε. 241. 241 πέρα της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 242 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε. 242. 242 παρακαλώ και Κλείνω το, την ψηφοφορία. Απερίφθη. 243. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να σηκώνετε τα χέρια όμως. Μη μας ταλαιπωρείτε. Αγαπητοί φίλοι. Ξέρω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ήτρε, αλλά τώρα ψηφίζουμε. Και λυπούμε δεν βλέπω στους αδέλφους που κάθονται εκεί πίσω. Ξαναρχίζω. 243 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύω. Πέρας. Απερίφθη. 244 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη με την ίδια πλειοψηφία 245 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 246 υπέρ Όχι, δεν πρέπει να ψηφίσουμε τη 246. Ζητώ συγγνώμη. 248 υπέρ. Κατά. Αποχές και επαληθεύω. 248. Πέρασε. Απερίφθη. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 257 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 258 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 262 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 10α υπέρ κατά αποχές. Έχουν και οι ε, πολιτικές ομάδες εσωτερικές ε, διαφοροποιήσεις. Να ψηφίζετε λοιπόν, να σηκώνετε τα χέρια. Συμβαστική 10. Δεκάλφα. και κλείνω την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 267 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 266 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 269 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 13 της NV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 της NV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 της NV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 274 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 275 υπέρ κατά επαληθεύουμε 275 πέρας της ψηφοφορία. Απερίφθη. 276 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 277 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 279 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 της ΕΝΒΗ υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 12 της ένβη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 15 της ένβη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 291 υπέρ. Κατά. Και επαληθεύουμε τη 291. 291 πέρας της ψηφοφορίας 293 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 294 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 19α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και επαληθεύουμε τη 19α, συμβαστική 19α. Επαλήθευση πέρα της προφορίας. Εγκρίνεται. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 297 υπέρ. Κατά αποχές. Επαληθεύουμε 297. 297 πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. 298 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική 19β υπέρ, 19β κατά αποχές. Εγκρίνεται 12 συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 δεύτερο τμήμα της ΕΝΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 303 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 56 της ΕΝΒ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 311 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απερίφθη αλλά σε παληθεύσουμε 311 Ένας υπεράριθμος από τους σοσιαλιστές δημοκράτες. Πέρας της ψηφοφορίες Και απερίφθη. 312 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 313 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 313 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 313 το δεύτερο τμήμα, έτσι. Πέρας. Ένας υπεράριθμος από τους σοσιαλιστές. Πέρας. Απερίφθη. 314 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 315 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 316 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 317 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 318 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 319 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 312 320 ε, υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε επαληθεύουμε 320 320 πέρας της προφορίας απερίφθη 321 υπέρ Κατά. Αποχές απερίφθη. 322 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 323 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 324 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 325 υπέρ κατά επαληθεύουμε 325 πέρας κύριε και θεέ απερίφθη 326 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 327 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 428 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ένβη 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένβη 46 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται, NV47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ένβι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά μάλλον απεριφθέλας επαληθεύσουμε την 19 επαληθεύουμε τη 19 πέρασε και απεριφθή μικρή διαφορά όμως 20 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 28 υπέρ, κατά απερίφθη, 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ, κατά αποχές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 Πέρας της 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για την τελική ψηφοφορία. Πέρας Εγκρίνεται λοιπόν με μία αποχή και πάω στην τελευταία ψηφοφορία. Όπως είχα ανακοινώσει... Θα πάμε τώρα στον κύριο Λεβαντόφσκι. On the preparation of the Προετοιμασία μετεκλογικής αναθεώρησης του MFF 2014-2020. Τροπολογία πρώτη υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 4 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές ε, απερίφθη συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά Αποχές απερίφθη 22 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 27 υπέρ. Κατά Επαληθεύουμε την 27 υπέρ. Ψηφίζουμε την 27 λοιπόν, να επαληθεύουμε. Πέρας, απερίφθη 28 υπέρ, κατά αποχές, απερίφθη 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τροπολογία 40 με προφορική. Αντιρρήσεις λοιπόν που ενδεχομένω να έχετε. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. 42 μαζί με την προφορική τροπολογία λοιπόν. Υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνονται. 42 υπέρ κατά αποχές και εγκρίνεται ηλεκτρονικά τελευταία ψηφοφορία για σήμερα ναι θα στεναχωρηθούμε που θα μας τελειώσουν οι ψηφοφορίες και εγκρίνεται και συγχαρητήρια συγχαρητήρια αγαπητοί συνάδελφοι και μείνετε μαζί μας μέχρι το 10.30 Okay. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. The today Dear uh, Κυρίες και κύριοι, θεωρητικά έχουμε στη διάθεσή μας 34 ε, λεπτά για τρία σημεία στην ημερήσια διάταξη. Ε, είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Στην Επιτροπή μας όλα είναι δυνατά, εάν οργανωθούμε καλά. Ξέρετε ότι πρόκειται για θέμα προς ε, πληροφόρηση καθαρά. Μπούζεκ, ε, Γκέρεκ και Φέντερλε. Αυτές, αυτά είναι τα τρία σημεία. Σας υπόσχομαι ότι θα μιλήσω μόνο πέντε λεπτά Πρόκειται για τον ε, προϋπολογισμό του 2017, εντολή για τον τριμερή διάλογο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τι συμπεριέλαβα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς. Αν θέλετε να μου πείτε κάτι, θα το δούμε εντάχει. Καταρχήν, ο προϋπολογισμός του 2017 πρέπει να περιέχει στοιχεία ανάπτυξης. Επίσης, ε, να βασιστούμε ε, στην γνώση η οποία θα πρέπει να μην αποκλείει κανέναν. Επίσης, για να φτάσουμε σε αυτή την ανάπτυξη, θα πρέπει να έχουμε πολυετή προγράμματα όπως COSME, ε, Horizon και ούτω καθεξής. Επίσης, θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τις γραμμές του προπολογισμού για τον ορίζοντα 2020 και το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Ως προς τον ε, ορίζοντα 2020 υπάρχει ε, ένας δείκτης επιτυχίας 13-14 ε, σε σχέση με το 2022 του 7ου προγράμματος. Άρα ο δείκτης επιτυχίας είναι πολύ χαμηλότερος. και υπάρχει ανεπαρκής χρηματοδότηση, ε, ιδιαίτερα ως προς την συνυπευθυνότητα και υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι στον ε, τομέα της έρευνας, στον ευρωπαϊκό τομέα έρευνας. Σημείο 4. Μίλησα για ε, επαρκή χρηματοδότηση για την ΕΝΙΖΑ, τον οργανισμό για την ασφάλεια της ε, πληροφόρησης, της μετάδοσης της πληροφόρησης. Θα μπορούσα να σας απαντήσω και ερωτήσεις αν έχετε θέματα. Σημείο υπαριθμό 5. Στον τομέα της ενέργειας που έχει μεγάλη σημασία, μετά θα σας μιλήσω και για το TTIP, θεωρούμε ότι η αποτελεί πρόκριμα για την ολοκλήρωση του τομέα της ενέργειας. Αυτό είναι απόλυτα σαφές αφορά την αποδοτικότητα και την ασφάλεια και, καθώς και την κοινή έρευνα. Και μας ενδιαφέρουν και τα κοινά σχέδια, ε, κοινού ενδιαφέροντος. Το σημείο παριθμών 6 της γνωμοδότησής μου μίλησα για επαρκή χρηματοδότηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, συνεργασία των ρυθμιστών στον τομέα της ενέργειας. Πρόκειται για τον οργανισμό Άσερ. Από τον Άσερ εξαρτώνται τα πάντα. Η ενέργεια, η εσωτερική αγορά, η ε, εποπτεία του συστήματος χονδρικής ε, πώλησης και ούτω καθεξής για το τομέα της ε, ενέργειας και βεβαίως και το κόστος διαβίβασης, το κόστος μεταφοράς. Όλα εξαρτώνται από τους ε, ρυθμιστές και τους οικονομικούς φορείς. Έχει μεγάλη σημασία η συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας. Και το 7 και το τελευταίο σημείο αφορά τα προγράμματα το πρόγραμμα ITER. Πρόγραμμα ITER και όχι ΙΤΡΕ. Υπάρχει μία μικροδιαφορά, χρειαζόμαστε υποστήριξη. Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολη υποστήριξη του προγράμματος ITER για τις νέες πηγές ενέργειας, αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσουμε την πορεία μας έτσι ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών. Επτά είναι τα σημεία λοιπόν. Αν έχετε ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Και αν έχετε και ε, υποδείξεις, ε, έχει καλώς. Ναι, έχετε το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ ε, σύντομος γιατί έχουμε και μεγάλο περιορισμό, χρονικό περιορισμό. Σας ε, ευχαριστώ για το ε, προσχέδιο αυτό, το οποίο μπορώ να δεχτώ ως βάση εργασίας. Θα ήθελα να τονίσω τρία σημεία τα οποία δεν πρέπει να αφήσουμε, να αφήσουμε κατά μέρος θα πρέπει να τα δούμε λεπτομερία. Οι επενδύσεις για την έρευνα και την καινοτομία είναι ζωτική σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, αλλά και για το μέλλον των δικτύων έρευνας και καινοτομίας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση ως προς τις ΜΜΕ δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τις κοινότοπες εκφράσεις ότι η ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε προγράμματα για τις ΜΜΕ, καθώς και τις νεοσύστατες εταιρείες και επιχειρήσεις. Το τρίτο σημείο είναι η επαρκής χρηματοδότηση που θα πρέπει να παρασχεθεί σε προγράμματα που θα επιτρέψουν την μετάβαση της οικονομίας μας, της κυκλικής οικονομίας που αποτελεί προτεραιότητα. Θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα στο εγγύς μέλλον. Δεν είναι μόνο ένα από τα θέματα κλειδιά είναι και ένας φορέας της ανάπτυξης. Αυτά είναι τρία στοιχεία που θα ήθελα να προσθέσω και συμφωνώ με το έργο σας. Για να απαντήσω άμεσα, λέει ο Πρόεδρος, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, για το υπαριθμόν ένα ζήτημα Ίσως θα πρέπει να πούμε κάτι περισσότερο, γιατί οι ΜΜΕ εντάσσονται στο κόσμο. Αυτός είναι ο πυρήνας εργασίας, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε και αυτή την ε, προσθήκη. Για την κυκλική οικονομία η ΕΜΒΗ είναι υπεύθυνη, όχι η Ήτρα, αλλά μπορούμε να προσθέσουμε και εμείς κάτι. Η ΕΜΒΗ λοιπόν κάτι θα συντάξει για την κυκλική οικονομία είναι πολύ σημαντικό και παραμένω ανοιχτό σε υποδείξεις. Συμφωνώ, Πρόεδρε, αλλά η κυκλική οικονομία θα πρέπει να έχει μία εξισορροπημένη θεώρηση και για τη διαχείριση των αποβλήτων και πρόκειται και για ένα σημαντικό βιομηχανικό τομέα και χαίρομαι ε, να συμπεριληφθεί αυτό το σημείο. Θα ε, θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μαραγκάλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εντάχει απλώς να πω ότι δέχομαι τα σημεία τα οποία εκφράσατε εκτός από το ίτερ όπου διαφωνούμε όπου ψηφίσαμε και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα λάβουμε υπόψη και την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για το ΙΤΕΡ. Και γι' αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί αυτό το θέμα στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. είναι ο πρώτος χρόνος μετά από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της προηγούμενης επταετίας. Θα δούμε τι θα γίνει μέσα στα πλαίσια της χρηματοδότησης, του χρηματοδοτικού πλαισίου. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ως τη στρατηγική μας ε, ε, διεύρυνσης ε, χρηματοοικονομικών μέσων έρευνα ορίζοντας 2020 και λεπτά. Και επειδή είμαστε στο πρώτο έτος μετά από τις συμφωνίες των Παρισίων θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα πρώτα βήματα για την για την πολιτική εφαρμογής ε, των αποφάσεων για τις κλιματικές αλλαγές. Να δούμε δηλαδή και άλλες δυνατότητες μέσα στα πλαίσια της βιομηχανικής πολιτικής. Και εδώ μιλάμε για αποδοτικότητα, ενεργειακή απόδοση, επενδύσεις και προγράμματα περιφερειακής σύγκλησης για να υπάρξει μείωση ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ευρώπης. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα να επεκταθούμε επί των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν ακούγεται ο Πρόεδρος. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ως προς το ελεκτικό συνέδριο το θέμα, το θέμα αυτό συζητήθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών Εβραίος, όπου συντάξαμε τη βασική γνωμοδότηση και λαμβάνω υπόψη ότι αυτή θα είναι και η βάση για τις αποφάσεις μας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχουν καθυστερήσεις πλέον σε σχέση με τις δαπάνες. Έχετε απόλυτο δίκιο σε σχέση με την ενδιάμεση αναθεώρηση και άλλα αποτελέσματα της συζήτησης, επιμηχανική πολιτική, αποδοτικότητα, συμφωνώ απόλυτα. Ο κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να εκφραστώ και εγώ. Όλοι συμφωνούμε ότι το 2014 χρωστούσαμε 25 εκατομμύρια ε, ως προς τους απλήρωτους λογαριασμούς και τώρα φτάσαμε στα 17 δις γιατί ε, ε, υπήρχαν, υπήρχε ανεπάρκεια ως προς τα σχέδια και τα προγράμματα. Και η Επιτροπή μέχρι σήμερα δεν έχει εκφραστεί ως προς τις επιπτώσεις της μη καταβολής της έλλειψης ε, πληρωμών, γιατί ξέρετε ότι οι πόλεις πρέπει να ε, πληρώσουν τους προμηθευτές και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρεβλώσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να μας δώσει μία ανάλυση των επιπτώσεων αυτών των ε, μη πληρωμών γιατί σε τρία χρόνια θα έχουμε ένα τέτοιο ε, νέο μεγάλο κύμα και εάν δεν ε, καταβάλουμε τις πληρωμές, τότε θα πρέπει να επομισθούμε τις συνέπειες. Γι' αυτό θα ήθελα η Επιτροπή να μας δώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Ναι, πράγματι, θα πρέπει να το προσθέσουμε στη γνωμοδότησή μας. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των μη καταβολών στον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα μαζί σας. Ο κύριος Μπενίτο Ζιλουάγκα. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Θα θέλαμε ο προϋπολογισμός, ο κοινοτικός προϋπολογισμός στον τομέα της ενέργειας να κατευθυνθεί στους στόχους των κλιματικών αλλαγών με βάση τη Συμφωνία των Παρισίων. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό ως προς την έρευνα, ιδιαίτερα στον ορίζοντα 2020, γιατί φέτος υπέστη περικοπές δυστυχώς. Και θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών μέσα στα πλαίσια του, της ενεργειακής πρόσμιξης, του ενεργειακού μείγματος. Ε, το επενδυτικό σχέδιο Juncker δεν κατάφερε να φτάσει σε υψηλές επενδύσεις, κάτι το οποίο θέτει να αμφιβόλο την πρόταση της Επιτροπής για περαιτέρω ε, χρηματοδότηση. Δεν υπήρξαν μεγάλες επενδύσεις, κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει και στο κόσμο για τις ΜΜΕ. Θα πρέπει επίσης να ε, υποστηρίξουμε, να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία σε περιφερειακό επίπεδο και τοπικό. Τέλος, σε σχέση με την χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ, όπως ήδη γνωρίζετε έχουμε αντιταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Θα πρέπει να σταματήσει η χρηματοδότηση αυτού του σχεδίου που αποτελεί μια μεγάλη μαύρη τρύπα στον τομέα της ενέργειας. Και κινούμαστε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή μιλάμε για ένα συγκεντρωτικό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται σε πολύ λίγα χέρια. Υπάρχει μεγάλη αμφιβολία ως προς την ασφάλεια και την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων και υπολοιμάτων. Γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσει το ίτερ κατά την άποψή μας. Ευχαριστώ. Συνάδελφε. Νομίζω ότι το θέμα της ενέργειας μαζί με το κλίμα θα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για τον ορίζοντα 2020, όμως θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο ορίζοντας 2020 ε, έχει κατά 40% υψηλότερη χρηματοδότηση από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. αλλά ε, ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, και μια πρόταση για περαιτέρω αύξηση προϋπολογισμού. Μιλάμε όμως για ένα 40% αύξηση. Ε, σε σχέση με το ίτερ μιλάμε όχι για τήξη, αλλά για σύνδεξη. Μιλάμε για σύνδεξη και γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και η βασική έρευνα. Η βασική έρευνα, η πρωτογενής δηλαδή έρευνα. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι το αμεληταίο, αλλά αυτό θα το δουν οι επιστήμονες. Η κυρία Κάπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, στην ουσία έχουν καλυφθεί τα θέματα. Πρόκειται για μια επαρκή χρηματοδότηση που ζητούμε και για το Horizon 2020 και για το Connecting Europe Facility. Το επισήμανατε και εσείς. Είναι κάπως χαμηλότερο το επίπεδο υλοποίησης σε σχέση ε, με το ΕΦΣΥ και νομίζω ότι θα πρέπει στην ενδιάμεση αναθεώρηση να την ενισχύσουμε. Και νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότησης. Ε, ίσως θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε εδώ όμως και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του κόσμου. Βεβαίως είναι σημαντικά όλα αυτά ε, για την ε, ένβη, αλλά θα πρέπει και εμείς να παρακολουθήσουμε το θέμα. το βασικό είναι να μην περικοπούν τα κονδύλια για να γυρίσω στο θέμα του λέει ο Πρόεδρος, αυτό που λέμε είναι «We want our money back». Θέλουμε πίσω τα λεφτά μας. Και μάλιστα όχι απλώς πίσω τα ίδια, αλλά δεκαπλάσια ζητάμε. Κόντιτσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα συμπληρώσω αυτό που είπε ο συνάδελφος Μάνκα. Ότι δηλαδή Πρέπει να πιέσουμε την Επιτροπή να αποκαταστήσει τα ποσά που χάθηκαν. Γιατί δεν μπορούν να εκτελεστούν οι πληρωμές, δεν μπορούμε να εξοφλήσουμε τους λογαριασμούς. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να το καταφέρουμε. Για δε το ΙΤΕΡ, Αυτό που δεν λέει ο συνάδελφος είναι ότι αυτά που, αναζη, ε, ερευνούνται μέσω του ΙΤΕΡ έχουν να κάνουν με την ηλιακή ενέργεια. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Κυρία Κάπελ, θέλετε πάλι το λόγο. Α, όχι, εντάξει. Uh, uh, και σα ευχαριστώ. Οι παρατηρήσει ήταν πάντα πολύ εύστοχε. Τι λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν και σα ευχαριστώ. Έχετε λοιπόν την προθεσμία για τις τροπολογίες. 24 Μαρίου ενδεικτικές προτάσεις για πιλωτικά προγράμματα 31 Μαΐου 12 τροπολογίες 24 6 το απόγευμα και ενδεικτικές προτάσεις για πιλωτικά έργα 31 12 το μεσημέρι και νομίζω ότι αυτά ήταν τα σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο για τη, με την Επιτροπή των Προπολογισμών Ασφαλώς. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ψήξη και τη θέρμανση με εισηγητή τον Άνταμ Γκίρεκ που παίρνει και το λόγο. Και ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω θα πρέπει να ακολουθήσω τη δική σας μέθοδο, Πρόεδρε. Ε, και και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Η στρατηγική για την ψήξη και τη θέρμανση αφορά τη χρήση περί του 40% πρωτογενούς ενέργειας. Έχει τεράστια σημασία ως θέμα, εκ των οποίων ε, το 50% είναι χρηστική ενέργεια και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με την αξιοποίηση, με την μετατροπή της ενέργειας σε θέρμανση ή ψήξη, ε, αν το συγκρίνουμε με την ηλεκτρική. Η παραγωγή λοιπόν ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί κατά κάποιο τρόπο να ενοποιηθεί στην αγορά ενέργειας ίσως, αλλά η ψήξη και η θέρμανση έχει πολύ πιο τοπικό χαρακτήρα με σημαντικά ζητήματα που πρέπει να επιλύονται σε τοπικό επίπεδο. Και πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι έτσι συμβάλλουμε σε μια διαφοροποιημένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων και δράσεων που θα πρέπει να λαμβάνονται τα μεγαλύτερα αποθέματα που αφορούν τα κράτη που εντάχθηκαν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004 έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό τον ενεργειακό των κτηρίων. Το ταχύτερο, η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική μέθοδος για την αποτελεσματική χρήση ενέργειας και ταυτόχρονα δημιουργεί και πολλές θέσεις εργασίας. Και γι' αυτό αυτός ο στόχος, αυτή η προτεραιότητα πρέπει να καλυφθεί με επαρκή πόρους, πρέπει να ε, καταρριφθούν τα ποσοτικά όρια στα, στο Περιφερειακό Ταμείο την περιφερειακή ανάπτυξη. Υπάρχει όριο λοιπόν, ε, ένα μεγάλο σφάλμα που θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, απαλληφθεί και αυτό σε σχέση με τα πεπαλαιωμένα κυρίως οικιακά συγκροτήματα, τα μεγάλα εκείνα συγκροτήματα της κομμουνιστικής εποχής. Πρέπει λοιπόν να στραφούμε προς την ε, αναμετατροπή των συγκροτημάτων και, την, ε, και κυρίως τη μετατροπή τους σε κέντρα ε, παραγωγής ενέργειας και συμπαραγωγής ενέργειας εδώ θα θυμίσω ότι είμαστε από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης σε, με μεγάλη, σε πολύ ψηλά επίπεδα κατανάλωσης ε, φυσικού αερίου. Αντίστοιχα στις περιοχές της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην ψήξη. Με μεγαλύτερη κατανάλωση λοιπόν ε, ηλεκτρικής ενέργειας που θα απαιτηθεί για την ψήξη για τα συστήματα ψήξης. Ε, όλα αυτά λοιπόν σημαίνουν πως χρειαζόμαστε επαρκή εργαλεία, σχεδιασμό, αρχιτεκτονική, χωροταξία, φυσικές πηγές, ε, θέρμανσης και ψήξης θα πρέπει να αξιοποιηθούν, θα πρέπει να ενισχυθεί η καινοτόμως ενέργεια και να εγκαθιδρυθεί ένας ολόκληρος κλάδος ε, παραγωγής, έρευνας και παραγωγής που θα τίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Και εδώ βεβαίως, όπως είπα, πρόκειται για ένα νέο κλάδο, μια νέα εξειδίκευση στην Ευρώπη που θα ε, μας επιτρέψει να διατηρήσουμε την πρωτοκαθεδρία μας παγκοσμίω. Υπάρχουν ζητήματα και θέλω να επισημάνω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 27 Μαΐου. Πολύ σύντομα δηλαδή και η ψηφοφορία ε, προβλέπεται για τις 12 Ιουλίου στην Επιτροπή μας. Ολομέλεια τον Αύγουστο. Και σας ευχαριστώ λέει ο μιλητής τον Αύγουστο, διότι από ό,τι γνωρίζουμε δεν προβλέπεται. Ε, το ΕΛΚ τώρα, σκιώδης Thank you, Chairman. Ε, I, can... Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ τον εισηγητή και συμφωνώ μαζί του το θέμα της ε, θέρμασης και της ψήξης είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένα σε διάφορους χώρους και πλαίσια. Για την συγκεκριμένη έκθεση να πω ότι φύγει πολλές σημαντικές τεχνικές πτυχές αλλά πιστεύω πως απαιτούνται περισσότερες στρατηγικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υποβληθούν τροπολογίες και θα θίξω κάποια σημεία προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να γίνει αυτή, η τοποποίηση. Υπάρχουν ε, διαφορετικά ζητήματα που αφορούν την ψήξη και τη θέρμανση ανάλογα με το κράτος και εδώ εμπλέκονται οι περιφερειακές κυβερνήσεις, ε, οι κοινότητες, οι δήμοι, όλα τα επίπεδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ενδυναμωθούν περαιτέρω, θα πρέπει να ε, ενθαρρύνουμε την ε, τεχνική ουδετερότητα, τεχνολογική ουδετερότητα. Πιστεύω ότι χρειάζεται να εξεταστεί το ζήτημα και περαιτέρω από οικονομικής πτυχής, οικονομικής πλευράς. Η θέρμανση και η ψήξη πρέπει να ειδωθεί στο πλαίσιο της ε, αλλαγής του κλίματος και οι διάφορες οδηγίες που αφορούν την ψήξη και τη θέρμανση και την ε, εφαρμογή αυτής θα πρέπει να είναι, μας δώσουν την βάση προκειμένου να ξέρουμε πού ακριβώς πάμε. Πρόεδρος, παρακαλώ είστε σύντομοι. Κύριος Πέτερσεν είναι απόνομος αγορητής, σκιώδης, συγητής από την Άλντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. και εμείς ε, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της θέρμανσης και ψήξης ε, αλλά και τα ζητήματα ασφάλειας ε, που ανέφερε ο συνάδελφος Άλακας. Η κρίση του αερίου πρόσφατα ήταν κρίση που οφείλεται στις θέματα ακριβώς της καλύτερης βελτίωσης της παράδοσης ε, αυτών των προϊόντων αερίου που έχουν και φυσικά επιπτώσεις στην δημιουργία θέσης απασχόλησης. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν θα πρέπει να είναι να δημιουργήσει το απαραίτητο ρυθμιστικό περιβάλλον και αυτό έχει τεράστια σημασία. Όπως επίσης και θέματα νομοθεσίας ε, για την ε, λειτουργία και κατασκευή των διαφόρων κτηρίων σε θέματα ψήφισης και ασφάλειας. Θα πρέπει να βρεθούν ολοκληρωμένες λύσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα και θα πρέπει να μπορεί να χορηγείται ε, ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα υποβάλω λοιπόν και εγώ και όπως και η ομάδα μου ε, τροπολογίες προς την κατεύθυνση και προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία με τον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρα. Ευχαριστώ συνάδελφε, σκιώδη ηγητής των Πρασίνων, ο κύριος Βάλεντε του απουσιάζει, ο κύριος Τούρμες βρίσκεται. Ευχαριστώ τον κύριο Γκίρεκ. Ε, ναι, χρειάζονται να γνωρίζουμε ότι τα ΕΦΣΙΣ δεν προβλέπουν πολλά προγράμματα για την ε, ροή χρημάτων προς την κατεύθυνση αυτή. Η HP είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προωθηθεί και να χρησιμοποιεί φυσικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιομάζα, ε, παίζει μεγάλο ρόλο στην ε, ψήξη και μια ερώτηση προς εσάς. Όταν λέτε ότι είστε υπέρ της τεχνολογικής ουδετερότητας, ο κύριος Γκίρεκ στην παράγραφο 15 αναφέρει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα πεπαλαιωμένε πεπαλαιωμένες καταστάσεις, Δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε άνθρακα στην, για την θέρμανση των ε, κατοικιών. Ειδικά για το θέμα της ε, θέρμανσης ε, νομίζω δεν είναι ο πιο σωστός τρόπος παροχής θέρμανσης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν νέες τεχνολογίες, να μην παραμείνουμε σε παλαιωμένε. Ευχαριστώ η κυρία Ένστ, προσωπεί την ΒΟΕ ως κοιοδησηγητρία. Σας ευχαριστώ. Στα περισσότερα θέματα πρέπει να πω ότι μας εξέπληξε θελτικά η έκθεση. Βεβαίω και εμεί πιστεύουμε ότι η αποτελεσματικότητα στη χρήση τη ενέργεια πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Και αυτό βέβαια στο χώρο του, ε, της ψήξης θέρμανσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ε, και οι ανανεώσιμε βέβαια πηγέ πρέπει να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο. Η έρευνα λοιπόν. Η έρευνα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως και το τονίζουμε αυτό. Τονίζουμε επίσης και το γεγονός ε, ότι έχουμε αντιμετωπίσει περικοπές στα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά. Και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση, μια τάση που δεν μπορούμε να δεχθούμε, μια τάση δηλαδή επιστροφής στα ορυκτά καύσιμα. Ε, πρέπει να δοθεί ε, ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα αυτά. Πρέπει να κοιτάξουμε το θέμα του υδραερίου, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να τονιστεί η σημασία των ανανεώσιμων πηγών, για να είναι σαφής η κατεύθυνση που επιδιώκουμε να ακολουθήσουμε. Τα παραδοσιακά ε, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας πρέπει να εγκαταλειφθούν σταδιακά ε, και νομίζω ότι γι' αυτό για να συστήσουμε για μια νέα στρατηγική για τέτοια σημαντικά ζητήματα θα έχει νόημα να προσδιοριστεί αυτή η σαφή τάση, αυτή η σαφή κατεύθυνση προς την οποία θέλουμε να προχωρήσουμε, τα ανανεώσιμα και βέβαια η ε, ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη χρήση της ενέργειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω των μέσων που έχουμε στη θέση μας. Πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά η αποτελεσματικότητα και πρέπει να πω ότι η αποτελεσματικότητα δεν έχει να κάνει καθόλου με, τον, με το παλαιό κομμουνιστικό σύστημα. Μετά την κατάρρευση του κομμουνιστικού συστήματος υπήρξαν κτίρια που χτίστηκαν χωρίς να έχουν προβλέψει την ενεργειακή αυτάρκεια ή αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας και σε αυτό θα πρέπει να γίνει σχετική προσαρμογή και σε αυτό πρέπει να είναι οι προσπαθίες μας. Ευχαριστώ. Ζητώ από τους διερμηνείς να παραμείνουν άλλα 10 λεπτά. Η κατάσταση δεν είναι συνήθις, δεν συμβαίνει συχνά. Θα φροντίσουμε λοιπόν να κλείσουμε τη συνεδρίαση 10 λεπτά αργότερα από τον προγραμματισμένο χρόνο. Επόμενος αγορητής είναι η κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη αναφέρθηκε το 50% της κατανάλωσης ενέργεια ε, χρησιμοποιείται στην θέρμανση και την ψήξη. Προκτεί λοιπόν για το μεγαλύτερο τομέα κατανάλωση ενέργειας και έχει πολύ μεγάλη σημασία ως εκ τούτου. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση σε τέσσερα σημεία τα οποία ήδη έχει επεξεργαστεί επαρκώς η έκθεση ε, η συγκράτηση της θερμικής ενέργειας, ιδιαίτερα βέβαια σε ε, σχέση και με το διοξείδιο του άνθρακα από τα κτίρια, η πιο αποτελεσματική χρήση της ενέργειας από τα κτίρια, όπως γνωρίζετε σε ένα πρόγραμμα REFIT ε, ε, μπορούν να προχωρήσουν αυτές οι προσαρμογές με χαμηλό κόστος Ε, θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί ο ρυθμός ε, προσαρμογής των ε, κτίριων που είναι πολύ χαμηλός αυτή τη στιγμή, είναι ακόμα 2%. σε σχέση με την χρήση της θερμικής και ψυκτικής ενέργειας. Ευφυή κτίρια, επίσης ένα άλλο σημείο, ευφυή κτίρια και ευφυή συστήματα ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση της ζήτησης. Για να γίνει αυτό ωστόσο χρειάζονται κονδύλια για την έρευνα ένα αριθμιστικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει και κίνητρα για την αξιοποίηση των σχετικών ε, πόρων, η παραγωγή ψυκτικής ενέργειας βεβαίως στις νότιες κυρίως χώρες και εδώ νομίζω μπορούμε να επιμείνουμε ιδιαίτερα στην καλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας και τελευταίο σημείο καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των ηλιακών εγκαταστάσεων ε, βασικά αποκεντρωμένη αξιοποίηση της ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα, επιμέρους ομιλητές. Ένα λεπτό καθένας. Κύριε Μπλάνκο Λόπες και μετά κύριε Κόλιτσεκ. Okay, Mr. ο κύριος Μπλάνκο Λόπε, ο κύριος Κόχλιτσεκ έχει το λόγο. Ενάμιση λεπτό λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να βρούμε ε, μία τεχνική υφής ε, λύση. Υπάρχει όμως μία πρώτη πτυχή που είναι πολύ σημαντική και αφορά τη στρατηγική. Πρόκειται για θεωρητικές μελέτες. Ε, στα, σε πανεπιστήμια στη Δρέσδη υπάρχει μία θεωρία που επιτρέπει την χρήση μίας συγκεκριμένης μονάδας για τη θέρμανση και για την ψήξη. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στις θεωρητικές αυτές μελέτες για το μέλλον. Έχουμε μία τεχνική λύση, αλλά υπάρχει και το θέμα των επιπτώσεων. Γιατί υπάρχουν επιπτώσεις ε, σε σχέση με την δημιουργία υδρατμών και θα πρέπει να δούμε ποια είναι και η επίδραση επί του ύδατος. Να δούμε δηλαδή αυτά τα δύο σημεία, οι θεωρητικές μελέτες και το θέμα των αποβλήτων να ληφθεί υπόψη από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκεται μαζί μας ε, ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Ντόνελη. Α, όχι, δεν είναι παρούσα η Διευθύντρια. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να μας πει λίγα λόγια για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε καταγράψει τα σχόλια της Επιτροπής και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η έκθεση, δηλαδή η τελική έκδοση της έκθεσης και θα δούμε τι δράση θα ακολουθήσουμε για τη θέρμανση και την ψήξη μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής μας. Δεν έχουμε χρόνο για να μιλήσω για τα επιμέρους σημεία, αλλά συμφωνούμε με αυτά που προελέχθησαν σε σχέση με την θεμελιώδη σημασία της ε, ενέργειας, της αποδοτικότητας της ενέργειας για την σωστή ψήξη και θέρμανση κτηρίων, τη μόνωσή τους και ούτω καθεξής. Πολύ χρήσιμα αυτά τα στοιχεία και περιμένουμε την ε, έκθεση στην τελική της μορφή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκίρεκ, ο εισηγητής, ε, ευχαριστώ πολύ. Εντάχει γιατί δεν έχουμε χρόνο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια μακρά συζήτηση επί του θέματος, αλλά από πλευράς τεχνικών ζητημάτων δεν γράφουμε τίποτα νέο στο έγγραφο. Ξέρουμε τι να χρησιμοποιήσουμε για τη θέρμανση ή την ψήξη ανάλογα ε, με το σε ποια χώρα βρισκόμαστε και τι διαθεσιμότητες έχει. Νομίζω όμως ότι στην γενική εικόνα θα πρέπει να ορίσουμε τις προτεραιότητές μας και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία στη συζήτηση με τους σκιώδεις. Θα δούμε τις προτεραιότητες αυτές όπως ορίζονται. Η μία από αυτές είναι η αναβάθμιση των κτηρίων γιατί δείτε τα κτίρια στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, πώς θέλετε να τα ε, μονώσετε. Υπάρχουν ε, πολλά παλιά κτίρια που χρειάζονται αυτή την ε, αναβάθμιση ως προς τη χρήση ενέργειας. Επίσης, από τις χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 υπάρχουν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα από τέτοια κτίρια, γιατί δεν έχει νόημα να ε, υπάρχει θέρμανση αν δεν υπάρχει σωστή μόνωση των κτίριων. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε έναν κατάλογο προτεραιοτήτων. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Άνταμ Γκέρεκ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω προθεσμία για τροπολογίες 27 Μαΐου 12 η ώρα και θα ψηφίσουμε στην Ήτρε στις 12 Ιουλίου και μάλλον το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώσαμε και με το σημείο υπαριθμών 12-13 τώρα. Οι οικονομικά ε, ε, αποδοτικές επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών και του αποτυπώματος του άνθρακα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ε, στον κύριο Φέντερλε και ιδιαίτερα τους Σκιώδης, γιατί δεν έχουμε χρόνο. δεν ε, μπορούμε να εξετάσουμε την έκθεσή σας. Μπορώ να προτείνω κάτι για το μέλλον. Καταρχήν ε, να αναβάλουμε τη συζήτηση στις 13-14 Ιουνίου, δηλαδή στην επόμενη συνάντηση της Ήτρε, σε τρεις εβδομάδες να αλλάξουμε βεβαίως και την προθεσμία υποβολής ε, τρυπολογιών για τις 15 ε, Ιουνίου μετά τη συνεδρίαση της ε, προσεχούς Ήτρε. Αυτή είναι η πρότασή μου. Δεν νομίζω ότι έχουμε και άλλες δυνατότητες. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή, τον κύριο λέει, να μας πει τι σκέφτεται για αυτή την κατάσταση, την πρόταση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για όποιον ήθελε να λάβει μέρος στη συζήτηση, ΜΚΟ, εμπλεκόμενος φορείς, κυβερνήσεις, μια από μεγάλη απογοήτευση, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Μπορούμε να έχουμε ε, μια σωστή συζήτηση σε σχέση με το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών. Θα πρέπει λοιπόν να ανακοινώσουμε το, το πότε θα διενεργηθεί η συζήτηση και βεβαίως η προθεσμία να μετατεθεί για μετά από την συζήτηση έτσι ώστε και το κοινό να μπορέσει να, το ευρύ κοινό να μπορέσει να συμμετάσχει. Ε, Λυπάμαι για τους συναδέλφους που περίμεναν αυτή τη συζήτηση, αλλά θα επανέλθουμε σε λίγες εβδομάδες και θα γίνει μια σωστή συζήτηση, όπως αρμόζει στο θέμα αυτό. Ευχαριστούμε, Φρεντερίκ. Θα πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και στο Στρασβούργο να έχουμε μία έκτακτη συνεδρίαση, αλλά σε αυτή την περίπτωση ε, ίσως άλλοι συμμετέχοντες να μην μπορέσουν, σημερινοί δηλαδή, συμμετέχοντες να μην μπορέσουν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση, μόνο διαδικτυακά να την παρακολουθήσουν. Μπορούμε να το σκεφτούμε και αυτό και θα δούμε ε, στο εγγύς μέλλον ποια είναι η καλύτερη λύση και θα έρθουμε σε επαφή με εσάς και εσείς μετά με τους υπόλοιπους σκιώδεις. Ζητώ συγγνώμη σε όλους που είχαν ετοιμαστεί για τη σημερινή συζήτηση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεδρίαση. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς, λέει ο πρόεδρος, μείναν 13 λεπτά παραπάνω. 13-14 Ιουνίου θα ξανασυνεδριάσουμε και ίσως ενδιάμεσα και στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ πολύ.